Σας ευχαριστώ. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα για τα μέλη των ε, Ευρωβουλευτών σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τη σύγκρουση των συμφερόντων, χθες, 15 Ιουλίου 2014, σχετικά με τα πέντε μέλη το, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ε, τα ονόμασα κανονικά μέλη. Σας ευχαριστώ για το χειροκρότημα, λέει ο Πρόεδρος. Uh -huh. Πρώτη φορά, πρώτη φορά με χειροκροτάτε. Uh Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, με ακούτε? Μάλιστα, πολύ ωραία. Ας ξαναξεκινήσω λοιπόν. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Συμπεριφορά ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τι ε, συγκρούσει οικονομικών συμφερόντων, χθε 15 Ιουλίου 2014, ε, ονόμασα και διόρισα τα πέντε μέλη της Επιτροπής. Δάνουτα Χούμπνερ, Μαντιντελβό Στέρες, Σαγιάτ Καρίμ, Φρανσίσκο Σουζαβάκνα και Ζέρι Μασταλικά. Είναι αναπληρωματικά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και θα διοριστούν τις επόμενες ε, ημέρες γιατί θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δεν έχουμε ακόμα λάβει οριστική απάντηση από όλους. Τα πέντε τακτικά μέλη μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν τις εργασίες του και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την προθυμία ε, και για τη συνεργασία τους. Ε, Κύριος Γκλέζος, ζήτησε διαδικαστικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, χθε το πρωί ο πρόεδρος Γιούγκερ δήλωσε ξεκινώντας την ομιλία του ότι τα όνειρα έχουν θέση εδώ. Ύστερα από λίγο τα όνειρα τουλάχιστον της δημοκρατίας καταστράφηκαν όταν αρνήθηκε ο αγαπητός πρόεδρος Σούλτς να δώσει το λόγο για να εξηγήσει ο συνάδελφος Παπαδάκης για ποιο λόγο δεν τον εκφράζει η Λεπέν. Ήταν ενός δευτερολέπτου εξήγηση και το αρνήθηκε. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί καταστροφή της έννοιας της δημοκρατίας και ζητώ από τον πρόεδρο Σούλτς, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά, να αναγνωρίσει το λάθος του. Σας ευχαριστώ κύριε Κλέζο. Στο κοινοβούλιο αυτό μπορεί να πάρει κανείς ε, το λόγο για να κάνει διαδικαστικό θέμα, όπως και εσείς. Έτσι, το λόγο για διαδικαστικό σας το έδωσα το λόγο, όχι για την ημερήσια διάταξη, ούτε για θέματα κανονισμού, αλλά μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Παπαδάκης δεν έκανε το ίδιο χθε. Ε, ξαναζήτησε το λόγο, μάλλον δεν ζήτησε το λόγο, ούτε ε, έκανε ε, κάποιο μήνυμα ότι ήθελε να μιλήσει. Και πήρε απλά το λόγο μπροστά από 750, 750 συναδέλφους. Αν πάρνει καθένα το λόγο έτσι, δεν υπάρχει δημοκρατία ούτε θα ξέρει και κανείς τι έχει πει ο άλλος. Και γι' αυτό λοιπόν παρακάλεσα τον κύριο Παπαδάκη να περιμένει και να ζητήσει κανονικά το λόγο. Και αν το είχε ζητήσει κανονικά θα τον είχα δώσει. Δεν ε, μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Πολύ απλά δεν γίνεται αυτό και κατά τα άλλα πρέπει να πω ότι έδωσα στον κύριο Παπαδάκη το λόγο και την ευκαιρία να εκφραστεί ως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και να πει ότι ως μία εγγυγραμμένος δεν εκπροσωπείται από την κυρία Μαρή Λεπέν. Αυτό το καταλαβαίνω και ε, το καταλαβαίνω δημόσια. Μίλησε εξ ονόματος των μη και όχι για δικό του λογαριασμό η κυρία Λεπέν. Νομίζω ότι είναι σαφές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στην διορισμό τεσσάρων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ έχουμε... Ε, ακούσαμε ότι υπάρχει ε, διαδικαστικό πάλι έτοιμα. Äh, Κυρία Χάρμς, ε, κύριε Σούλτς, κύριε Πρόεδρε, για μας ε, πιστεύουμε ότι σε ό,τι αφορά την πρόταση για το μεταβατικό αυτό στάδιο ε,